Ο κύριος πρόεδρος. ευχαριστώ. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε λέει ο πρόεδρος, συνάδελφε, αρχίζουμε. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση η οποία είχε διακοπεί στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν, άρα τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Έχω δύο ανακοινώσεις για το σώμα.